μας βοήθησε να προσχωρήσουμε στην ενιαία αγορά. Θα επαγρυπνούμε για να δουλέψουμε στο θέμα αυτό και να συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες δομές που είναι αναγκαίες. Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις ψήφου. Διακόπτουμε μέχρι τις 3. señor presidente. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι.